102 μάλλον, ε, όπου παρουσιάζεται ότι έχει εγκριθεί 40 βουλευτές πρέπει να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους μέσα σε 48 ώρες. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε εγκρίνεται. Αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν με ακούει τόσο ή άλλως ό,τι και να λέω.